και εφόσον πρόκειται για ένα σημείο πάρτιμά μας ήδη και ο ιδιοκτήτης ε, έλυσε και το θέμα του ε, ενοικίου του επομένου, της επομένης ριετίας και θα λύσουμε και το πρόβλημα του αμιάντου. ο ιδιοκτήτης έχει δεσμευτεί ότι ε, όσες μονώσεις δεν, δεν είναι ασφαλείς έναντι ε, του αμοιάντου θα διορθωθούν και αυτό μας ενδιαφέρει διότι διαφορετικά θα έπρεπε να κάνουμε ούτως ή άλλως επενδύσεις ε, για κλιματιστικά, για πυρασφάλεια ε, και αν δούμε άλλωστε τις τουαλέτες των συνεργατών μας δεν είναι και λαμπρές άρα πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που δεν έχει αναβαθμίσει ο ε, ιδιοκτήτης ε, ε, τα τελευταία χρόνια αλλά πρόκειται για ένα κτίριο που δεν είναι εγκαταλελειμμένο είναι χτισμένο απλούστατα εδώ και 80 χρόνια οπότε εγώ που ασχολούμαι χρόνια με τα κτίρια πρέπει να πω ότι χρημαζόμαστε μία σύντομη προοπτική ε, και ε, το κτίριο Ρεμάρ ε, τέθηκε προς συζήτηση την τελευταία στιγμή. Πρέπει λοιπόν να πω ότι είμαστε λιγάκι απογοητευμένοι που μας ειδοποιήσατε τόσο πρόσφατα. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει η μεταφορά το Δεκέμβριο και να μην την αφήσουμε για τον, τις αρχές του έτους όπου θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Οπότε είμαι υπέρ αυτής της αγοράς. Ωραία. Ευχαριστώ. Ε, εάν οι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις ε, θα τους έλεγα να τις θέσουν να απαντήσει μια και καλή ο Γενικός Γραμματέας διαφορετικά του δίνω το λόγο κατευθείαν ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λέει ο Γενικός Γραμματέας ε, όσον αφορά τη, τα κτίρια πρέπει να σας πω ότι μπορώ να προσπαθήσω να αναφερθώ στις ε, μεταφορές πιστώσεων για το τέλος του χρόνου διότι για το 2010 είχαμε πει να καταρτήσουμε ένα απόθεμα 11 ε, εκατομμυρίων το οποίο διαθέτουμε ακόμη και να έχουμε κατόπιν αποφάσεως της Προεδρίας ε, επιπλέον 5 εκατομμύρια τα οποία έχουμε άρα αυτά τα ποσά μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν. 24 Μαρτίου αποφάσισε το Προεδρία μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια και για την πληροφορική. Ήταν ε, μία από καιρού επιθυμία της Επιτροπής Προϋπολογισμού, δηλαδή να μην εξετάζουμε ένα κτίριο μετά το άλλο, αλλά να έχουμε μία στρατηγική πολιετή η οποία βαθμία θα εφαρμόζεται. Και πιστεύω ότι στα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό ότι το κτίριο Ρεμάρα αναφέρεται ήδη στην παράγραφο 33 της στρατηγικής κτιρίων του Μαρτίου σαν πρόθεση αγοράς. Έτσι έχει εντοπιστεί ε, έπρεπε να βρεθούν οι πόροι αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα έγγραφο το οποίο μας ενδιαφέρει από καιρού διότι ήδη έχει ενταχθεί στα κτίρια μας και όπως είπε και η κυρία Χολμάγερ ε, δεν είναι ένα κτίριο που πρέπει να έχει κανείς πρόσβαση από έξω αλλά είναι άμεσα σε, σύνδεση με το έθριο των ε, δύο άλλων κτιρίων. Ε, όσον αφορά την στρατηγική κτηρίων βλέπουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνται όλα τα κτίρια μας γεωγραφικά ώστε να μην χρειάζεται να οργανώνουμε και μεταφορές από το ένα κτίριο στο άλλο και επιπλέον ισχύει και το ρητό καλύτερα να αγοράζουμε παρά να νοικιάζουμε ε, ε, ήδη έχουμε αγοράσει το 83% των εκτάσεων που καταλαμβάνουμε και δεδομένης της ε, χρηματικής κατάστασης ε, θα θέλαμε να εξοικονομήσουμε τα ενίκια. Γι' αυτό και το κτίριο Ρεμάρ τώρα το οποίο έχει 8.500 τετραγωνικά μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο στην στρατηγική μας κτηρίων για να την ολοκληρώσουμε τα ποσά τα οποία υπολείπονται ε, πέραν των 11 εκατομμυρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διότι έχουμε εξοικονομήσεις από το ενεργειακό κόστος με μείωση της ε, κατανάλωσης ενεργείας και σε ορισμένα σημεία ε, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το 2011 οπότε όσον αφορά τους πόρους για τα κτίρια έχουμε ορισμένα παρόλο που θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια για αυτή την αγορά περισσότερα από ό,τι είχαμε αρχικά προϋπολογίσει. Όσον αφορά το Wi-Fi ε, είχαμε προβλέψει προτεραιότητες για τα προγράμματα του Προεδρίου και η μεσοπρόθεσμη στρατηγική η οποία αποφασίστηκε στις 23 Μαρτίου του 2010 υπήρχε ένα θέμα 2 Β Connectivity and Wi-Fi όπου λέγεται σαφώς ότι έχουμε την φιλοδοξία να αναπτωρισόμεθα με όλο και πιο ευέλικτες ε, και ε, κινητές επικοινωνίες ε, και στους χώρους εργασίας και στα γραφεία των Ευρωβουλευτών να υπάρχει δηλαδή η μεγαλύτερη δυνατή επέκταση Οπότε τα 5 εκατομμύρια που είχαν ε, προβλεφθεί γι' αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα από το Προεδρείο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 εκατομμύρια από τα προβίζολα από απροπιέωσεων και 800.000 από τις temporary allowances για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου. Βεβαίως υπάρχουν και ε, οι προδιαγραφές ασχαλείας οι οποίες πρέπει να γίνονται γίνονται σεβαστές και για τους εσωτερικούς χρήστες και για τους εξωτερικούς χρήστες παρόλο που οι μεν και οι δε έχουν διαφορετικά δικαιώματα προσβάσεως πρέπει όλοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ε, τη χρήση του διαδικτύου, το Wi-Fi. Υπάρχουν βέβαια ακόμη ορισμένα σημεία ασαφή, ε, τι θα γίνει με το γραφείο γραφείο της Σόφιας το ποσό εκεί είναι κάτω από τα 10 εκατομμύρια υπάρχουν διαπραγματεύσεις δεν μπορώ ακόμη να σας πω ακριβώς περί τίνος πρόκειται αλλά υποθέτω ότι το ποσό το οποίο να αναφέρουμε ε, είναι περίπου 9 εκατομμύρια και αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί και ε, η επιθυμία να αγοραστεί ήδη αναφέρεται εις ε, τη στρατηγική των κτηρίων στον αριθμό 38. Έχουμε άλλωστε και ένα βασικό σημείο ασάφειας πριν από το τέλος του χρόνου, δηλαδή πότε ε, θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις προσαρμογές των μισθών, ε, διότι ε, αν απορριφθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορισμένα ποσά τα οποία δεν έχουν περιληφθεί ή στον προϋπολογισμό θα πρέπει να συνυπολογιστούν και θα χρειαστεί ε, να ε, προβλέψουμε 8,3 εκατομμύρια επιπλέον αλλά αυτό που έχει σημασία δεν ε, είναι πότε θα ληφθεί η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με, ε, το, με την ακύρωση της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά πότε θα αποφασίσει για το νέο ποσοστό αυξήσεως των μισθών πράγμα το οποίο ίσως δεν γίνει ε, φέτος και θα ισχύσει πλέον από το 2011 εάν όμως γίνει ακόμη το Δεκέμβριο και ε, βγει αυτή η απόφαση και πρέπει να γίνουν αυτές οι πληρωμές μπορώ να σας πω ότι θα κάνουμε οικονομίες σε άλλες γραμμές του υπολογισμού που αναφέρονται στο προσωπικό και θα μπορέσουν να καλύψουν αυτό το ποσό. Το σημασία έχει πότε θα αποφασίσει το Συμβούλιο, αλλά έχουμε ε, προβλέψει και τις δύο εναλλακτικέ, δηλαδή είτε γρήγορα οπότε θα έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις πληρωμών το 2010 και αν υπάρχει μεταφορά στο 2011 θα δημιουργηθούν ορισμένα περιθώρια και αντιλαμβάνουμε ότι και στις τωρινές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2010 τα σημεία αυτά είναι σημαντικά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 Εάν υπάρξουν και άλλα περιθώρια τότε φαντάζομαι ότι ίσως θα μπορέσει κανείς να κάνει και άλλες επενδύσεις για την τεχνολογία ε, ε, στο διαδίκτυο ε, διότι αυτό που έχει σημασία για τους βουλευτές είναι να είναι καλά εξοπλισμένοι και ιδίως οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές του 2009 πιστεύουν ότι έχουν να καλύψουν κάποια διαφορά. Δηλαδή αν χρειαστούν επενδύσεις θα ήταν καλό να μπορέσουμε να τις καλύψουμε και πιστεύω ότι θα το χαιρέτιζαν πολλοί ευρωβουλευτές. Εάν βρούμε τη σχετική στήριξη για τα μέτρα αυτά τότε πιστεύω ότι συνολικά θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά νομίζω ότι βρισκόμαστε σε, σε ένα επίπεδο εκτελέσεων στο 98% υπάρχουν ορισμένες ασάφειες διότι τώρα είναι δυνατόν εις την γραμματεία ε, να μεταφέρουν ορισμένα ποσά στο επόμενο έτος και δεν ξέρουμε στο παρελθόν πόσο έχει γίνει αυτό και πόσα δηλαδή χρηματικά μέσα έχουν διατεθεί. Θα σας μπορέσω να σας το πω αργότερα αυτό καλύτερα από ό,τι σήμερα, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν ορισμένες επενδύσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εκτελέσουμε σωστά το προϋπολογισμό μας. Ευχαριστούμε το Γενικό Γραμματέα για αυτήν την διεξοδικότατη ενημέρωση ε, για την συνεπέστατη περιγραφή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για φέτος και για το ε, πρόγραμμα αγοράς του ακινήτου ΓΝΑΧ. Ο κύριος Βόγκε έχει ζητήσει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ. Θα πω κάποια πράγματα εντάχει και για τα δύο ζητήματα. Ε, εξ τον του Βλαντιμίρ που είναι εισηγητής αλλά δεν μπόρεσε να παραστεί η σημερινή συνεδρίαση για την αγορά του κτηρίου Ραμάρ. Ο κύριος Μάγκη, ο ε, δέχεται την αγορά του ακινήτου και δέχεται την, ε, ε, τη μεταφορά πιστώσεων για τους λόγους που εξέθεσε η κυρία Χολμάγερα και ο Γενικός Γραμματέας. Η εγκύτητα του κτηρίου, η διαθεσιμότητά του, η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης, η ιονία απώλεια του κτηρίου από άλλο αγοραστή, αν δεν κινηθούμε γρήγορα, ε, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Ε, ο εισηγητή θα κάνει και κάποια σχόλια νομίζω για τη διαδικασία που καλό θα ήταν να τα έχει κατά νου και ο Γενικό Γραμματέα πρώτον για το δημοσιονομικό κανονισμό ε, το Κοινοβούλιο έχει δύο εβδομάδες ε, για να αποφασίσει αν θα εκδώσει γνωμοδότηση. Στην έκθεση σωστά αναγράφεται ότι δεν επαρκούν ε, οι δύο εβδομάδες και προτείνεται παράταση σε οχτώ εβδομάδες και νομίζω ότι θα υπάρξει γενικότερη υποστήριξη για αυτή την πρόταση επίσης. Ε, για την κτηριακή πολιτική του Κοινοβουλίου. Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες στην αρχή του έτους, αλλά ε, στο τέλος του 2010 τελικά ακόμη δεν έχουμε εκδώσει γνωμοδότηση για την αγορά κτηρίου, οπότε μάλλον αυτό ε, υποδεικνύει ότι δεν είναι σωστή η στρατηγική μας. Καλό θα ήταν ίσως να αναθεωρηθεί. Ελπίζω ο Γενικός Γραμματέας να δεχτεί την αγορά και τη μεταφορά. Δεύτερον, για τη διεύρυνση της πρόσβασης με σύρματο δίκτυο στο, στις και στο Στρασβούργο αναγνωρίζεται σίγουρα ότι έχουν γίνει ήδη προσπάθειες και το Προεδρείο έχει προσπογράψει την πρόταση και μάλιστα θα συμφωνήσετε ότι είναι καλό να διευρύνουμε το ασύρματο δίκτυο σε όλα τα κτίρια, εάν ε, ε, είναι δυνατόν αυτό. Είμαστε από τα λίγα βασικά θεσμικά όργανα της Ένωσης όπου τα κτίρια δεν έχουν ε, πλήρη πρόσβαση πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, σύνδεση στο διαδίκτυο. Ε, κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Πρώτον, ε, είναι χαλεπή η κυρία από οικονομικής πλευράς. Ε, κάναμε δυσχερέστατες οικονομικές συζητήσεις με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό και συνεχίζονται και θα τεθούν ερωτήματα. Μπορούμε τώρα να δώσουμε 4 εκατομμύρια για να διευρύνουμε το, την κάλυψη του ασύρματο δικτύου στο Στρασβούργο, ενώ λίγες μέρες το μήνα επισκεφτόμαστε αυτό το κτίριο. Ε, ε, επίσης, υψηλό κόστος, 7,5 εκατομμύρια ευρώ 4 εκατομμύρια, εκ των οποίων είναι για το Στρασβούργο. Φαίνεται υψηλό αυτό το κόστος. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να αιτιολογήσει αυτό το υψηλό κόστος ή να κάνει ένα επιμερισμό ε, του, του κόστους, γιατί δεν νομίζω να είναι τόσο περίπλοκη η τεχνολογία ε, του ασύρματου δικτύου. 7,5 εκατομμύρια για δύο κτίρια μου φαίνεται ένα υψηλό πόσο ο εισηγητής προτείνει να, να υποστηρίξουμε τη διεύρυνση του εισκάλυψη του ασύρματου δικτύου στις Βρύξε. Βρυξέλλες, αλλά δεν δέχεται τα 4 εκατομμύρια για την επέκταση στο Στρασβούργο ε, και νομίζω ότι η τελική του θέση θα είναι συνάρτηση των απαντήσεων που θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας Ευελπιστός σε ερωτήσεις που έκανα. Ευχαριστώ από συνάδελφοι, η Έλγα Τρίπελ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την λεπτομερή ενημέρωση και να σας πω ότι η αγορά του κτηρίου Ρεμάρ μας βρίσκει σύμφωνους με τον τρόπο με τον οποίο ε, παρουσιάσατε τα διάφορα στοιχεία. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα κτίρια στις Βερξέλλες ε, θεωρώ ότι είναι σωστά τα πράγματα. Αντιθέτως συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν για το Στρασβούργο είναι προφανές. Ε, πρέπει πάντοτε να δούμε τι επενδύσεις μπορούν να αιτιολογηθούν ε, ανα πάσα δεδομένη στιγμή. Όσον αφορά το κόστος προσωπικού και πότε πρόκειται να υπάρξει ε, απόφαση του δικαστηρίου. Είπατε κύριε Γενική Γραμματέα ότι αν χρειαστεί να διαθέσουμε ακόμη ποσά το 2010 είναι 2,8% 2,8 εκατομμύρια ευρώ και ε, θα προέλθουν από εξοικονομήσεις. Πρόκειται ε, για από ποιον τομέα που έχετε εξοικονομήσει. Δεν το κατάλαβα πολύ καλά και θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα κάτι για το σύρματο δίκτυο. I would like to ask you something, Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, Γενική Γραμματέα. Για, το, για τη διαδικασία, για την κάλυψη του ασυρμάτου δικτύου και τις προτάσεις που κάνατε. Ε, σίγουρα δεν είμαι ο μόνος. Όλοι θέλουμε να έχουμε σύγχρονες τεχνολογίες και το ασύρματο δίκτυο σε όλα τα κτίρια. Όμως, βλέποντας την πρότασή σας, λέτε εσείς ότι θα έχουμε την ε, πιο προηγουμένη τελευταία γενιά τεχνολογίας, ε, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα για την ταχύτητα και την αξιοπιστία του δικτύου. Όμως δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και βλέπω και τα ποσά. 4 εκατομμύρια περίπου για τα κτίρια στο Στρασβούργο και 4 περίπου για τις ε, Βρυξέλλες. Φαίνεται μάλλον υψηλό το κόστος. Έχετε δημόσιο ασύρματο δίκτυο σε πολλά μέρη, έτσι, σε δημόσιους χώρους, σε πολλές πόλεις. Ε, και οι τιμέ αναφορέ είναι κατά πολύ χαμηλότερε. Ποια είναι αυτή η προηγμένη τεχνολογία που είναι τόσο ακριβή. Ε, ε δηλαδή, η ε, τελικά αξίζει να δαπανίσουμε τόσο πολλά χρήματα για αυτή την τεχνολογία. Ευχαριστούμε κύριο Φινάντης, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα για την ενδελεχή τοποθέτησή του, για την εκτηριακή πολιτική. Συμφωνούμε ε, με την πολιτική, συμφωνούμε με την αγορά του κτηρίου. Για, ε, για το Wi-Fi, για το ασύρματο δίκτυο. Δεν έχει νόημα να έχουμε δίκτυα ασύρματα στις Βρυξέλλες ε, και να μην έχουμε στο Στρασβούργο. Άρα συμφωνούμε να επεκταθεί το ασύρματο δίκτυο σε όλους τους χώρους εργασίας μας. Σίγουρα είναι ένας τρόπος για να γίνουμε κι εμείς πιο αποδοτικοί και να εργαστούμε εξυπηρετώντας το στόχο της νομοθετικής αριστείας. Ε, επιβεβαιώνουμε ότι έχουν όλοι εργαστεί αποτελεσματικά και σίγουρα είναι το χαμηλότερο δυνατό κόστος για να έχουμε αυτή την προηγμένη τεχνολογία και για τα, την ταχύτητά τη και για την ανάλυση κόστους, ωφέλου, όλα αυτά τα στοιχεία που ζήτησαν οι συνάδελφοι, σίγουρα θα μα τα δώσει ο Γενικός Γραμματέα. Δεν έχουμε καθόλου ενστάσει ούτε για το θέμα του ασύρματου δικτύου, ούτε για την κτηριακή πολιτική. Ο Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η Μόνικα Χολμάιερ ζήτησε το λόγο. Να ακούσουμε πρώτα το Γενικό Γραμματέα ή θέλετε το λόγο πριν, μετά θέλετε. Πολύ ωραία. Ο γενικό Γραμματέας. Ευχαριστώ. Καταρχήν σας ευχαριστώ διότι υπάρχει ευρία στήριξη σχετικά με το κτίριο Ρεμάρ και οι ερωτήσεις που ετέθησαν αναφέρθηκαν στην ε, ασύρματη επικοινωνία και ε, σε άλλα δαπάνες. Ε, επίσης υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επενδύσουμε στο Στρασβούργο γιατί περνούμε εκεί αρκετό χρόνο και ακόμη ακόμη πιο σημαντικό διότι οι συνθήκες εργασίας στο Στρασβούργο είναι πολύ περίπλοκες, έχουμε μικρά γραφεία, ελάχιστες μόνιμες δομές και πρέπει να μπορούμε να έχουμε πιο ευέλικτες τεχνολογίες πληροφόρησης και εδώ είναι πιο οξύ το θέμα από ό,τι στις Βρυξέλλες και γι' αυτό το Προεδρείο αποφάσισε παρόλο που χρησιμοποιούμε λίγο στο Στρασβούργο ε, το Στρασβούργο να βελτιώσει τις ε, υπηρεσίες που προσφέρονται και στο σημείο αυτό. Οι ε, περικοπές κόστους προέρχονται από μία μελέτη η οποία έγινε και η οποία υπευλήθη εις το Προεδρείο. Η κυρία Τρίπελ έκανε μία συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τα 8,2 εκατομμύρια, δηλαδή που εξοικονομεί αυξήθηκαν τα 8,2 εκατομμύρια και που μειώσαμε τις δαπάνες προσωπικού. Στον τομέα του προσωπικού αυτή τη στιγμή μέχρι ε, ε, το τέλος του 2010 ε, έχουμε μειώσει στους μισθούς 4,4 εκατομμύρια στο σημείο 200 υπόλοιποι υπηρεσίες 1,2% και στις αποστολές ε, εξοικονόμηση 2,4 εκατομμύρια. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε εξοικονομήσει 11 εκατομμύρια και μπορούμε να πούμε ότι ακόμη και αν χρειαστεί να ε, αυξήσουμε τις δαπάνες μας ε, σε αυτό το επίπεδο θα έχουμε περισσότερα να διαθέσουμε για τις δαπάνες προσωπικού από αυτά που θα μας ζητήσει το δικαστήριο. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια η Μόνικα. Ε, ευχαριστώ. Όσον αφορά το Wi-Fi, την ασύρματη επικοινωνία, ε, για μας ε, είναι πολύ δυσάρεστο ότι τα κτίρια του Κοινοβουλίου μένουν άδεια τόσο καιρό γιατί δεν μπορούμε να εργαστούμε σωστά. Δηλαδή, εάν θέλετε, ε, αν θέλετε να παρακολουθήσετε μία συζήτηση εκτός του γραφείου σας είστε περιορισμένος, δεν έχετε χώρο. Οπότε υπάρχει μία αίτηση από 300 βουλευτές να υπάρχει Wi-Fi στους χώρους που εργάζονται και δεν πρέπει να τσακωνόμαστε τη στιγμή που δεν έχουμε ε, στενότητα πόρων. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και ε, ε, οι συνάδελφοι οι οποίοι υπέγραψαν τον το, την αίτηση αυτή είναι ε, διακομματική. Ε, θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να μπορεί κανείς να συμμετέχει στο κοινοβούλιο σε μία συζήτηση χωρίς να ε, μιλάει και να μπορεί να δουλεύει και αυτό ισχύει για όλα τα σημεία όπου εργαζόμαστε να, δυνα... να μπορούμε να έχουμε επικοινωνίες και συνθήκες εργασίας καλές. Είναι ε, κάτι ε, το οποίο ε, συνεπάγεται στη σύγχρονη εποχή. Έχω και άλλα σχόλια, να τα πω τώρα ή αργότερα. Τώρα, τώρα, λέει ο πρόεδρος. Ωραία. Σχετικά με το ε, έγγραφο εργασίας το οποίο έχω καταρτήσει θα ήθελα να σας πω ότι αναφανώς ήθελα με αυτόν τον τρόπο να ε, ε, ενημερώσω τους συναδέλφους για τη γενική κατάσταση και επίσης να αναφερθώ και στην δημοσιονομική, στον δημοσιονομικό κανονισμό διότι εδώ δεν είναι πολιτική κάθε θεσμικό όργανο καλύπτει τα δικά του συμφέροντα εκτός από τα γραφεία πληροφόρησης. Εν τω μεταξύ έχει γίνει κάποια πρόοδος στο επίπεδο αριθμών αλλά εάν προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε ε, ποια κτίρια έχουν ποια αξία τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα διότι οι αριθμοί απέχουν πολύ ε, ε, και αυτό γιατί γιατί δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία άλλοι συμπεριλαμβάνουν κάνουν το θεωρητικό ενίκιο, άλλοι υπολογίζουν τα πάρκινγκ και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα έπρεπε μία φορά να συμφωνήσουμε σε μία σύντομη ε, ε, ε, κατάταξη των αριθμών η οποία να είναι διαφανή γιατί κάποιος που ασχολείται με αριθμούς έχει δυσκολία να ρίξει μια ματιά και να μπορέσει να αποκομίσει μια εντύπωση του τι συνεπάγονται όλοι αυτοί οι αριθμοί και αυτό μπορεί να σας το πω εν ονόματι όλων των συναδέλφων. Εν τω μεταξύ έχουμε και μία στρατηγική αγορών υπό τον όρο ότι η αγορά είναι πιο συμφέρουσα από το ενίκιο ή το leasing ε, με τη λογική ότι έχουμε περισσότερο συμφέρον. Ε, εν τω μεταξύ όμως Βλέπουμε ότι η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να ξέρουμε αν εκεί χρησιμοποιούν άλλες προδιαγραφές και γι' αυτό κάνουν περισσότερα leasing και περισσότερες ενοικιάσεις. Όσον αφορά την, ε, τους, ε, τις δημόσιες προκηρύξεις διαγωνισμών για τα κτίρια, για το έγγραφο Ρεμάρ δεν μπορούσαμε να κάνουμε προκήρυξη διαγωνισμού, έπρεπε να αποφασίσουμε το θέλουμε ή όχι. Αλλά παλαιότερα έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ των τρόπων χρηματοδότησης των οποίων διαθέταμε διότι δεν είχαμε μέσω πρόθεσμη δυνατότητα χρηματοδότησης διότι ο προπολογισμό ήταν ετήσιος και δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε ε, δάνεια και γι' αυτό οι διαδικασίες στο παρελθόν ήταν διαφορετικές. Τώρα και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση αυτή αλλά για το fitting out ποτέ δεν έχει γίνει προκήρυξη διαγωνισμού διότι εάν νοικιάζουμε τότε αναλαμβάνει ο, ο ιδιοκτήτης ε, ενώ αν αγοράσουμε η κατάσταση είναι διαφορετική. Τώρα, όσον αφορά ε, τις οι ειδικέ κατασκευές χρηματοδοτήσεως. Ε, δηλαδή είτε μαζεύουμε ε, ποσά από το ραμασάζ το Δεκέμβριο ή προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε και πιο νωρίς ό,τι διατίθεται αλλά καλό θα ήταν να έχουμε μία, ένα πρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό και εδώ αναφέρομαι εις ε, το ΚΑΤ που μέχρι πρότινος ήταν πολύ ενδιαφέρον αλλά ε, το θέμα είναι ότι ε, προσπαθούμε να έχουμε σε ένα κτίριο όλους τους 3.000 υπαλλήλου χωρίς να τους χωρίζουμε σε 7 κτίρια ε, τα οποία μας κοστίζουν ετησίε 27 εκατομμύρια άρα βλέπετε ότι δεν θα εξοικονομήσουμε και λίγα άρα σημασία δεν έχει ε, να, να νοικιάζουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβά. Όταν βεβαίως συζητάμε για τις προδιαγραφές του Λουξεμβούργου το καταλαβαίνω αλλά δεν έχουμε επιλογές αυτή τη στιγμή διότι εφόσον έχουμε 3.000 υπαλλήλου εκεί πρέπει κάπου να τους εγκαταστήσουμε αποτελεσματικά και αξιοπρεπώς. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η εξέλιξη είναι θετική και βέβαια πιστεύω ότι και στο μέλλον δεν θα έχουμε ποτέ αποθεματικά πολύ μεγάλα. Αυτό που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι η δημοσιονομική αρχή στο ε, ενημερώνεται την τελευταία στιγμή για την πολιτική κτηρίων. Δεν υπάρχει μία μακροπρόθεσμη προοπτική και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στις 8 εβδομάδες οι οποίες αναφέρθηκαν και δεύτερον να σας πω ότι καλό θα ήταν να ενημερωνόμαστε εγκαίρως όταν ξεκινά κάποιος να προγραμματίζει κάτι διότι θα ήθελα να ξέρω τι θα γινόταν αν υπήρχε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο θα κόστινε ε, στις ε, εκατομμύρια και 8 εβδομάδες πριν θα λέγαμε ε, δεν μας αρέσει όλα θα είχαν εντωμεταξύ προετοιμαστεί, θα είχαν προκηρυχθεί, θα είχαμε εξοδέψει ένα σωρό λεφτά οπότε δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε στο τέλος να λαμβάνουμε αποφάσεις γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει μία κλιμακωτή διαδικασία ή στη δημοσιονομική διαδικασία κατά τρόπον ώστε σε καταρχήν να ενημερωνόμαστε, να επηρεάζουμε και στη συνέχεια να συνοδεύουμε και να παρακολουθούμε το κάθε πρόγραμμα. Διότι υπάρχουν εντωμεταξύ και συγκριτικές τιμές της αγοράς, διότι πολλές φορές λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λεφτά και μπορούν να πληρώσουν φουσκωμένες τιμές. Αυτό δεν πρέπει να ισχύσει και θα πρέπει το Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα να συνεργάζονται για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο. Στο έγγραφο γίνονται πολλές ερωτήσεις προς τα θεσμικά όργανα και θα ήθελα κάποια στιγμή σε μερικούς μήνες να το ξανασυζητήσουμε στην ημερησία διάταξη για να μας απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πώς διαβλέπουν δηλαδή το μέλλον διότι θεωρώ ότι αυτό είναι και αναγκαίο και λογικό πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο τελευταίες ερωτήσεις γιατί μετά έχουμε και ψηφοφορία κύριοι και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Βόμπη. Για τις δύο μεταφορές. Είπα και πριν ότι δέχομαι την πρώτη γιατί φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ των συναδέλφων, αλλά πιο δύσκολη είναι η περίπτωση για το Wi-Fi, όπου είπε ο Γενικός να εγκρίνουμε τη μεταφορά, αλλά όχι για το Στρασβούργο, για μας αυτό είναι δύσκολο. Ζήτησα από τον Γενικό να μας κάνει μια κατανομή του κόστους. Πολλοί είχαν πει ότι είναι πολλά τα 7,5 εκατομμύρια και παρακαλώ να αναβληθεί η ψηφοφορία μέχρι να μας δοθεί η κατανομή από τον Γενικό. Ευχαριστώ. Γκρέσλερ. Λοιπόν, ουσιαστικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μόνικα Χολμάγερ. Το, ενδιαφέ... το... έγγραφό της είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι εδώ και έξι χρόνια δεν ε, ε, είχα δει ένα έγγραφο το οποίο να παρουσιάζει την κατάσταση και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο. Όσον αφορά το Λουξεμβούργο, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να μας εξηγήσει ε, την κατάσταση διότι ασχέτως το τι προβλέπουν οι συνθήκες βλέπω ότι έχουν χτίσει 685 εκατομμύρια σε τιμές του 1980 οπότε υπάρχει μία άνεση αντιμετώπιση ήθελα λοιπόν να σας πω ότι τα δύο μεγάλα εργοτάξια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λειτουργούν τελείως διαφορετικά όσον αφορά το πρόγραμμα της Rue de la έχουμε επιφυλαχθεί και όσον αφορά αφορά το Νότο όπου πρόκειται να χτιστούν 250.000 τετραγωνικά μας λέγουν ότι είναι φτηνότερα αν όλα συγκεντρωθούν. Θα ήθελα όμως κάποιος να μου πει τι κερδίζουμε με το να χτίζουμε καινούργια κτίρια. Δηλαδή όλα αυτά θα ήθελα να τα ακούσω πιο προσεκτικά και πιο επιμελώς. Οι ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι γίνεται με τα δύο μεγάλα εργοτάξια στη και πότε θα ε, ισοφαρίσουμε ε, διότι κάποια στιγμή μας στέλνουν το λογαριασμό και μας λένε ότι τώρα μας κοστίζουν όλα πολύ λιγότερο από ό,τι είχαν προβλέψει. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα και τον Ισηγητή και όλους τους συνάδελφους που μίλησαν στη σημαντική αυτή συζήτηση τώρα. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που θίχθηκαν για το έγγραφο προς την Κομισιόν. Όσο δε για τις δύο μεταφορές, απαντάω στον κύριο Βόγγεν αμέσω. νομικά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε σήμερα τη μεταφορά γάμα 11 για το wi δηλαδή. Μπορούμε να το αναβάλουμε για την επόμενη φορά. Και εντωμεταξύ θα ζητήσουμε από το Γενικό Γραμματέα την κατανομή που ζητήσατε μεταξύ των τόπων εργασίας. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν σήμερα τη μεταφορά γάμα 11. Αλλά για το κτίριο Ρεμάρ και την εφαρμογή του 179 για την πολιτική των κτηρίων τίθεται το ερώτημα εάν γνωμοδοτούμε. Ο εισηγητής μας δεν θέλει, για τους λόγους που εξήγησε η εισηγήτριά μας μάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμφωνεί να μην γνωμοδοτήσει. Συμφωνείτε όλοι και όλες να μην γνωμοδοτήσουμε. Ομόφωνα. Δεν γνωμοδοτούμε. Άρα εγκρίνουμε την πρόταση του κυρίου Γενικού ο οποίος μας ευχαριστεί και εκείνος δεόντος. Τώρα η μεταφορά 10, όχι 11, αλλά 10. Χρηματοδότηση για την αγορά του Ρεμάρ. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής. Σας ευχαριστώ κατά. Ευχαριστώ αγαπητές. Ομόφωνη έγκριση. Λογικό, λογικό. Το 11 αναβάλλεται. Και τώρα, τελευταίο σημείο, η περίφημη μεταφορά 53 της Κομισιόν. Χαμηλά τα ποσά, 1 δισεκατομμύριο 500 εκατομμύρια. Και ο κύριος Σουριάν θα μας εξηγήσει περί τίνος πυρόκειται. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ. Δεν υπάρχει. Μπορούμε να δεχτούμε και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορώ να επαναλάβω ακόμη μία φορά ότι η Κομισιόν αύξησε στον τίτλο 1β σημαντικά τα ποσά πάνω από ένα δισεκατομμύριο μεταφέρεται εκεί. Τώρα, γιατί δεν ψηφίσαμε το πρωί μαζί με τις υπόλοιπες μεταφορές. Γιατί ο διορθωτικός 10 είναι σχεδόν τμήμα της μεταφοράς αυτής, αλλά όπως είπατε και εσείς θα ψηφίσουμε τον διορθωτικό προβλησμό 10 το Δεκέμβριο. Η μεταφορά όμως αυτή χρειάζεται για να μπορέσει να συνεχιστεί η δουλειά της Κομισιόν και δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην υποστηρίξουμε τη μεταφορά τώρα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Καμία απορία. Όχι. Βλέπω εδώ αντίχειρες προς τα επάνω. Ποιο είναι υπέρ της μεταφοράς αυτής που προτείνει η συγκήτρια. Ευχαριστώ κατά. Και εγκρίνεται η μεταφορά. Άψογα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδελφέ. Νομίζω ότι αν δεν απατώμε τελειώσαμε τη σημερινή μας συνεδρία. Η επόμενη θα γίνει στις 18. Στις 18 τι ώρα όμως. Ε, στις 18 στα 15 η ώρα. Μέχρι τότε πολλοί από εμά θα δραστηριοποιηθούν ιδιαιτέρως όπως η κυρία Ντουρό. Ιδιαίτερα όσοι και όσες είναι μέλη της αντιπροσωπείας για τη συνδιαλλαγή πρέπει να είναι διαθέσιμοι αύριο. Όλοι είμαστε διαθέσιμοι αύριο γιατί τη μήνυ ολομέλεια. Ιδιαιτέρως όμως γιατί στις 5, εκτός αν υπάρξουν αλλαγές, στις 5 θα συνεδριάσει ολόκληρη η αντιπροσωπεία για να αποφασίσει τη στρατηγική της στη συνδιαλλαγή που θα γίνει την 5η. Την 5η και ζήτησα ρητά να γίνει μετά την ψηφοφορία της Ολομέλειας. Ενώ δεν προβλεπόταν στην αρχή έτσι. Άρα μάλλον οι ψηφοφορίες της 5ης θα γίνουν στις 10 πιο νωρί. Αν όχι, τότε ως συνήθως στις 11 και τότε θα αρχίσουμε εμείς αργότερα. Κατά μία ώρα. Σας ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση. Λύεται.